Um, Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Για να ξεκινήσουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση. Προϋπολογισμοί και οικονομική με πολύ σημαντικά καθήκοντα σήμερα. Να ψηφίσουμε και να εγκρίνουμε το πρόγραμμα InvestEU. Πρώτα όμως Πρέπει να γίνει παρουσίαση των τροπολογιών. Πριν περάσω όμως αυτό, ας εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, αν δεν έχετε αντιρρήσεις. Ανακοινώσεις δεν έχω. Ας περάσω λοιπόν στην παρουσίαση των τροπολογιών. Όπως ξέρετε έχουμε εργαστεί εντατικά και ευχαριστώ και όλους τους κοιόδης για την ε, συμβολή στην προετοιμασία των συμβαστικών τροπολογιών. Και παρακαλώ τον Ζωζέ Μανουέλ να πει δύο λόγια. Και θα συνεχίσω κι εγώ. Δεν ξέρω αν κύριε και συμπρόεδρε με το δικό μου το μικρόφωνο θέλετε να πείτε κάτι. Κύριος Γκάιερ. Ναι, ζητώ συγγνώμη, εγώ φταίω που δεν ξεκινήσαμε λίγο πιο νωρίς. Γιατί κανένα από τα μικρόφωνα δεξιά δεν δουλεύει, εκτός από του Ρομπέρτο. Ίσως να μην δουλεύει και κανένα τα δικά σας. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι έπρεπε να περιμένουμε μέχρι να τελειώσει και τον καφέ του ο Ρομπέρτο για να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Αυτά. Μπορώ βέβαια να τα πω και από εδώ, αλλά ίσως καλύτερο ο Ρομπέρτο. Ναι, κερδίζουμε και χρόνο Ξέρουμε ότι υπάρχει δυσκολία στην άφηξη ορισμένων και έτσι για αυτούς κερδίζουμε χρόνο, περιμένουμε δηλαδή να φτάσουν. Ας γίνει όμως πρώτα αυτή η σύντομη ανταλλαγή απόψε, Ζωζέ Μανουέλ. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ. Και θα μιλήσω πορτογαλικά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον συνεισηγητή μας, κύριο Γκουαλτιέρη, για μια καλή συμβιβαστική λύση. μια εξαιρετική επιστολή και τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε μέσα σε αυτή την ε, ε, βουλευτική περίοδο το ζήτημα. Βέβαια, πάντα υπό την επιφύλαξη της έγκρισης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το δικό μας όμως κομμάτι της δουλειάς το κάναμε και κλείσαμε το φάκελο. Πέραν ότι των ε, κομματιών εκείνων και των ποσών που θα ορίσει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ελπίζουμε να δείξει την ίδια ετοιμότητα και το Συμβούλιο για εξέβρεση συμβαστικών λύσεων και σημείων πρόοδου σε έναν τομέα σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί χρειαζόμαστε πάντα επενδύσεις, χρειάζομαι πάντα μια Ευρώπη ανταγωνιστική, μια Ευρώπη η οποία δεν θα αποκλείει κανέναν, μια Ευρώπη όπου θα εξακολουθεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο η συνοχή, μια Ευρώπη που χρειάζονται οι επενδύσεις και για να λειτουργεί η αγορά και για να εξασφαλιστεί σε όρους γεωγραφικούς αλλά και θεματικούς ε, μια ισορροπία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ τον Ρομπέρτο αλλά και όλους τους άλλους συναδέλφους που συνέβαλαν στην διατύπωση, ε, διαμόρφωση αυτών των συμβαστικών τροπολογιών που έχουμε. Έλαβαν μέρος λοιπόν ε, όλες οι ομάδες. Ευχαριστώ Ρίτα, τον συνεισηγητή μου και τους σκιώδης για την υποστήριξη και τη συμβολή τον Οτμαρκάρα, στον κύριο Σάβαλη, ιδιαίτερος θα ήθελα να τους μνημονεύσω, καθώς ε, ενεπλάκησαν εντατικά στην ε, επεξεργασία του θέματος αυτού. Αλλά και πάλι τονίζω όλοι οι συνάδελφοι, οι σκιώδεις, αξίζουν ευχαριστηρίων. Έχουμε 30 μέσα επιπλέον του έτσε και θα ήθελα να πω ότι αυτό που προτείνουμε εδώ δεν συνιστά παράταση του έτσε του σχεδίου Juncker. Όχι. Εδώ έχουμε αξιοποιήσει το, το life, τα κονδύλια του life, ε, περιβαλλοντικά κονδύλια, ε, οτιδήποτε έχουμε δυνατότητα να αξιοποιήσουμε σε δημοσιονομικά προγράμματα μέχρι το 2020 και είναι απαραίτητο εν προκειμένου να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς τη λειτουργία της συμπληρωματικότητας στις υποδομές. Ιδιαίτερα και για τα κοινωνικά και για τα δημοσιονομικά μέσα τα οποία αφορούν το κοινωνικό ταμείο. Ε, ήμασταν πολύ προσεκτικοί βεβαίως στην διατύπωση των προτάσεων και τον προσδορισμό των στόχων που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των, ε, του Ταμείου Εγγυήσεων για την περίοδο μετά το 2021 δεν μπορούμε να μειώσουμε δηλαδή, δεν μπορούν να μειωθούν οι εγγυήσει και γι' αυτό έτσι ξέρουμε ότι θα έχουμε 38 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο αυτή ένα ποσό το οποίο έχει εγκριθεί στην Ολομέλεια, είναι άλλωστε σύμφωνο με τις θέσεις του Κοινοβουλίου για το Πολιετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και έτσι εδώ τώρα ενσωματώνεται η πρόταση αυτή στην έκθεσή μας. Η δε ψηφοφορία που έχει να κάνει με, ε, ε, το ποσό των εγγύσεων είναι μία ψηφοφορία που, δεν, ε, που έχει εξίσου μεγάλη συνάφεια με τα θέματα και τα ποσά του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου. Έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ποσά και για τις ε, μικρότερες επιχειρήσεις. Πόσο λεφτά έχω ακόμα, Πρόεδρε? Δύο λεπτά. Δύο λεπτά, όχι, όχι παραπάνω παρακαλώ. Καλώς πρόεδρε. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει το 75%, οι λοιποί πόροι θα αντιστοιχούν στο 25%. Πρέπει όμως πάντα να έχουμε μια ευελιξία σε σχέση με το συνολικό ε, ποσό της εγγύησης και ταυτόχρονα χρειάζεται και προβλεψιμότητα. και είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιηθεί και ε, η μέθοδος επιμερισμού μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το προσέξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σουζέ Μανουέλ, αξιότιμοι συνάδελφοι. Βλέπετε ότι αποκαταστάθηκε η τεχνολογία, είναι υπό έλεγχο. Συμφωνήσαμε με τον Ρομπέρτο Κουαλτιέρη να συντονίσω εγώ τη συζήτηση και στη συνέχεια ο Ρομπέρτο ε, να διευθύνει την ψηφοφορία. Ωραία. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Καλτιέρη, συνεισηγητή για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον συνεισηγητή Ζωζέ Μανουέλ Φερνάνδης, όλους τους και οδησηγητές και το προσωπικό και τους υπαλλήλους. Πολύ καλή συλλογική δουλειά. Οι συμβαστικές τροπολογίες έχουν εκπονηθεί με συνεργασία όλων των πολιτικών ομάδων και τα βασικά στοιχεία που θέλαμε να συμπεριλάβουμε είναι να ορίσουμε ε, το στόχο του policy window. Δηλαδή, όπως είπε και ο Σοζέ Μανουέλ, το πρόγραμμα αυτό συγκεντρώνει και συνενώνει διάφορα μέσα ε, χρηματοδοτικά και από τη μια θα πρέπει να έχουμε την αποτελεσματικότητα του ενιαίου ταμείου χωρίς να χάνουμε τις ε, ιδιαιτερότητες ε, των διαφόρων μέσων που συγχωνεύονται. Βελτιώνουμε τη διακυβέρνηση με το Διοικητικό Συμβούλιο και με καλύτερη σύνθεση του Συμβουλευτικού, Συμβουλευτικής Επιτροπής, διευκρινίζουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γραμματείας και βρήκαμε και μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους άλλους ε, φορείς που ασχολούνται με την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών. Υπάρχει και κάποια ευελιξία αλλά και κοινοβουλευτικός έλεγχος εξασφαλίζεται στη διαχείριση ε, της ε, ευελιξίας και της κατανομής μεταξύ των διαφόρων ε, παραθύρων ή θηρίδων. Και σε κάποια αιτιολογική σκέψη επίση διευκρινίζουμε και προσπαθούμε να επανεξισορροπήσουμε το γεγονός ότι έχουμε ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής τώρα στο Invest e και η παλιά όμως ε, αρχή της προσθετικότητας ε, δεν μπορεί ε, ούτε να χαθεί ούτε να επεκταθεί παντού. Γίνεται λόγος για την πολιτική ανεξαρτησία, για τον προσανατολισμό στην αγορά κτλ. Για να ληφθούν υπόψη οι διάφορες πτυχές και οι διάφορες απόψεις. Γενικά λοιπόν νομίζω ότι ήταν επιτυχία. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδης. Εμείς προσπαθήσαμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ανοιχτοί και δεκτικοί και ελπίζω να έχουμε μια καλή ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μας πιέζει λίγο χρόνος. Ευτό θα παρακαλούσα τους ομιλητές να τηρούν το χρόνο τους. Έχουμε προβλέψει τους και για ένα λεπτό. Δεν βλέπω τον κύριο Κάρας, έχει έρθει η κυρία Γαρδιά Σάμπαλ, η Αίντερ. Ας ψηφίσουμε τώρα, τι να πω, θέλω να ευχαριστήσω μόνο τους εισηγητές. Η τελική συμφωνία είναι καλή και ελπίζουμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο να μην αλλοιωθεί. Γιατί αυτό το σχέδιο επενδύσεων είναι καλό εργαλείο για να ξαναβάλουμε μπρος την ευρωπαϊκή οικονομία και να πετύχουμε τους βιώσιμού στόχους. Πολύ σύντομη. Ε, ο κύριος Πακέτα από το ECR. Να συγχαρώ του συνεισηγητέ για την εργασία που έκαναν στο θέμα αυτό. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έκαναν πολύ καλή δουλειά. Αλλά για εμά του κοιότε συνεισηγητέ, προφανώ ε, και εμεί δεν είχαμε αρκετό χρόνο. Αλλά προφανώ θέλαμε να προετοιμαστούμε για τον τριμερή διάλογο το συντομότερο δυνατόν. Θα προτιμούσαμε να είχαμε πιο πολύ χρόνο. Σε θέματα περιεχομένου, από πλευρά ECR υποστηρίζουμε την ιδέα του InvestEU. Έχει πολύ νόημα να συγχωνευτούν τα 14 αυτά ε, χρηματοδοτικά εργαλεία και γενικά μα ικανοποιούν οι συμβιβασμοί. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα τα είχαμε κάνει διαφορετικά, αλλά το κείμενο στο σύνολό του είναι αποδεκτό. Θα τονίσω μόνο τρία σημεία, με επιτρέπετε. Πιστεύω ότι το InvestEU θα αυξήσει τον αντίκτυπο στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και άρα δεν υποστηρίζουμε το συμβιβασμό για τον προπολογισμό. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πιο πολλά με πιο λίγου πόρου. Στην αρχική πρόταση η το θέμα της διαχείρισης ήταν πολύ περίπλοκο, αλλά πιστεύουμε ότι το κείμενο έχει βελτιωθεί πολύ. Θα προτιμούσαμε το EAB. η ΕΤΕΠ να είχε αναλάβει την διαχείριση κινδύνου και στην ε, όλη εγγύηση, όπως γίνεται στο ΕΦΣΥ, για να υπάρχουν και κάποιες διατάξεις ε, για την ε, Τράπεζα Επενδύσεων να αποφύγει και τη σύγκρουση συμφερόντων. Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι που όσοι είναι εταίροι εκτός ΕΤΕΠ θα έχουν πρόσβαση στον συμβιβασμό μας θα υπάρχει πλήρη πρόσβαση όταν θα μπει αυτή η δίκλυδα ασφαλεία. Αυτό αποτελεί μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τον ΕΦΣΥ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο κύριος Γκάιερ. Και χαίρομαι που έχουμε πολλούς προέδρους, που έχουμε πολλούς συναδέλφους που καταφθάνουν και αυτούς που νόμιζαν ότι ξεκινάμε στις 9. Καλώς ορίσατε. Καλημέρα. Ο κύριος Καράς, ο κύριος Μπαλτσέης έχει το λόγο από την Άλτα. Δεν είναι εδώ. Ο κύριος Τόρβαλτς. Ευχαριστώ. Να προσπαθήσω να τονίσω κάποια από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Με ένα χρονοδιάγραμμα όπως αυτό, η βοήθεια από τους βοηθούς και από τους συμβούλους είναι ανεκτήμητη και δεν είναι μόνο από τους δικούς μου βοηθούς ε, και, όλους τους, και με τους δικούς μου συμβούλους, από όλους τους συμβούλους. Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Να τονίσω τώρα κάποιες από τις προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη νέα δομή και τα, τις νέες ε, τράπεζες, τις εθνικές τράπεζες πρόθεσης. Βρισκόμαστε λίγο σε αχαρτογράφητα ύδατα. Είναι λοιπόν σωστή αυτή η απόφαση. Αντιμετωπίσουμε τις μεθόδους ε, εκτίμησης κινδύνου με σωστό τρόπο, δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για αλλαγές. Δεύτερο θέμα. Δομές. Δομές των διάφορων οργανισμών διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα σε ό,τι αφορά τη βελτίωση και τη διόρθωση των ζητημάτων. Τρίτο σχόλιο σε ό,τι αφορά τα τμήματα για τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό θα λειτουργήσει σε βάθος χρόνου. Όταν δε μιλάμε για τους λόγους αποτυχίας των αγορών, λόγους λέω αποτυχίας αγορών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτηματικά, πολλά εκκρεμή ζητήματα που οδηγούν στην αποτυχία της αγοράς. Δεν είναι μόνο η αγορά δηλαδή κατά αυτή η οποία από ό,τι χάνει. Ύστερα, το λέω και το ξαναλέω, έχουμε λίγο την τάση να φορτώνουμε λίγο το χριστουγεννιάτικο δέντρο με ευχές. Κύριε Τόρβαλτς, σας παρακαλώ να συντομεύετε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αυτά λοιπόν ήταν τα βασικά στοιχεία που είχα να σχολιάσω τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τρεμόσα. Κύριε Τρεμόσα. Herr Κύριε Τρεμόσα. thank you. I'm full... Ε, στα αγγλικά. Με κάλυψε απολύτως ο συνάδελφος Νίλ Στόρβαλτς και μπορούμε να προχωρήσουμε. Να επιταχύνουμε τη συζήτηση. Α, και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Ο κύριος Γίγκολτ από τους Πρεσίνους, παρακαλώ. Ε, ε, ο Ζόρντι θα τα πει πιο γρήγορα για τους Πρεσίνους. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ο κύριος Σολέ, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές και όλους όσοι εργάστηκαν στο θέμα αυτό για τη δουλειά που έκαναν. Για μας το σημαντικότερο ποιο είναι για τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεράσουμε αυτό το επενδυτικό έλλειμμα. Το αποφασιστικό είναι το κατά πόσο θα είναι πιο βιώσιμες αυτές οι επενδύσεις και από οικονομικής άποψης και από οικολογικής και περιβαλλοντικής. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να βελτιωθεί η βιωσιμότητα και η αηφορία, η καθοδήγηση προς τα εκεί και να επεκταθεί σε όλες τις ε, δράσεις και τις πολιτικές και τους στόχους δαπανών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το σχετικό κονδύλι είναι 65% και χαιρόμαστε που μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε και μια διάταξη για ανακαίνιση κτίριων βιώσιμη και με ενεργειακή απόδοση. Επίσης, αναφέραμε τη, αναφερέσαμε μάλλον την ε, αναφορά στην άμυνα, συμπεριλάβαμε μια αναφορά στην κοινωνική οικονομία, ε, στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και να προωθήσουμε γενικά την ισότητα, τη συμπεριλήψη διάστασης του, του φύλου και την περιφερειακή ε, ανάπτυξη, μάλλον τις περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες βέβαια δεν εξαιρούνται ρητά κάποια έργα που μπορεί να βλάπτουν το περιβάλλον. Έχουμε και κάποιες άλλες ανησυχίες, αλλά επειδή δεν έχω χρόνο θα πω ότι γενικά συμφωνούμε με τις συμβαστικές προτάσεις και ε, με τη θέση του Κοινοβουλίου που τελικά θα προκύψει από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω τον κύριο Παπαδημούλη ούτε την κυρία Ριάντα. Ο κύριος Βάλλη επίση αποσιάζει από το FTD. Η κυρία Κάπελ από το ΕΝΕΦ. E Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαστε ικανοποιημένοι, εγώ, με τους συμβιβασμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα InvestEU, γιατί έχουμε επενδυτικό έλλειμμα στην Ευρώπη από την ε, περίοδο της κρίσης και ελπίζω να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα Είχαμε και το έψη το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Τώρα να δούμε τι θα γίνει στην πράξη. Αν μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα ληφθεί υπόψη και να είναι πραγματικά μόνιμη αυτή η υπέρβαση του λίματος. Η μόχλευση είναι μεγάλη και όπως ήταν και στο ΕΦΣΙ και γενικά είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το εργαλείο και το ορίζω. Ähm, Ευχαριστώ. Μήπως κάποιος άλλος συνάδελφος της Επιτροπής να θέλει να λάβει το λόγο. Τώρα θα παρακαλέσω και για μας τους δύο έναν κατάλογο ψηφοφοριών, να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε. Για τους δυο μας εδώ, ένα κατάλογο. Κύριε Παπαδημούλη, να σας δώσω το λόγο. Παρακαλώ, εάν θέλετε βέβαια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω αυτές τις ώρες όλοι έχουμε μια πίεση λόγω της καθυστέρησης στα δρομολόγια για τους λόγους που γνωρίζετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συνεισηγητές για την προσπάθειά τους να έχουμε μια λειτουργική πρόταση και για το γεγονός ότι συμπεριέλαβαν αρκετές από τις προτάσεις μας. Το σχέδιο έκθεσης που θα κληθούμε να ψηφίσουμε αύριο έχει κάποια θετικά στοιχεία όπως η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, η στρατηγική για την Ευρώπη 2020, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, καθώς και η Οικονομική, Κοινωνική και Περιφερειακή Συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ, να, δεν μπορώ να συνεχίσω την ομιλία μου αν δεν επιβάλλετε κάποια ησυχία. Sie haben völlig recht, Herr Papa... Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παπαδημούλη, και ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ, παρακαλώ, αγαπητοί συναδελφοί. Ησυχία, ένδειξη σεβασμού προ τον ομιλούντα. Παρακαλώ. Το μικρόφωνο του ομιλητή, παρακαλούμε. But now you should use a Επισημαίνει επίσης τις διατάξεις για τις φυσικές καταστροφές, την προστασία του περιβάλλοντος και τα θέματα ενέργειας καθώς και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση μεταξύ άλλων στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική ευημερία. Πιστεύω ότι το ζήτημα των περιφερειακών ανισοτήτων απαιτεί μεγαλύτερη ανησυχία και πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην έκθεσή μας βάσει των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την εμπειρία των προηγούμενων δημοσιονομικών πλαισίων συμπεριλαμβανομένου και του EFSI το InvestEU αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δείξει εάν πραγματικά έχει ισχυρή πολιτική βούληση και προτεραιότητες για τη μείωση των ανισοτήτων κοινωνικών και περιφερειακών. Μπορεί να γίνει ένα εργαλείο που να ενισχύσει τις περιφέρειες και τους τομείς εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη αποεπένδυση τα τελευταία χρόνια. Να βοηθήσει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να καταπολεμήσει ισχυρότερα την ανεργία, να βοηθήσει στην ένταξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Τα θέματα της διαφάνειας και της λογοδοσίας είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικά και πιστεύω ότι έχουν γίνει κάποια μικρά, έστω ανεπαρκή βήματα σε αυτή την έκθεση. Η αιτήσια υποβολή εκθέσεων και αναφορών από τα όργανα του InvestEU, της EIB και της Επιτροπής είναι απολύτως απαραίτητα για τη δημοκρατική λογοδοσία. Όσον αφορά στα τέσσερα παράθυρα, κατανοούμε τη σημασία όλων τους και καλωσορίζουμε την πρόβλεψη. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι διατηρούμε αρκετές επιφυλάξεις στο σύνολο της έκθεσης, γι' αυτό και δεν θα την υπερψηφίσουμε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να στεί κανείς άλλο στο λόγο. Και έτσι προτείνω να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες και παρακαλώ τον Ρομπέρτο Κουαλτιέρη, συμπρόεδρο, να αναλάβει. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε νομίζω να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Εκτός και αν ο κύριος Βάλλη θέλει κάτι όχι. Κάνουμε πρώτα μια δοκιμαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Αρχίζει. Α, όχι, όχι. Περιμένουμε τρία ακριβώς λεπτά γιατί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες πριν τις 9 και 15. Όχι. Α, δεν το έχουμε γράψει πουθενά ότι στις 9 και 4 θα ξεκινήσουμε και έτσι μπερδευτούν οι συνάδελφοι. 10. 9. Α, ε, εντάξει. Το αποσύρω λοιπόν. Κάναμε και τη δοκιμή μας. Καλωσορίζω και την κυρία Βίλμπερν από τους σοσιαλιστές. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ και αρχίζουμε με το, η ψηφοφορία στο InvestEU. Ε, κάναμε τη δοκιμά μας όπως είπαμε και αρχίζουμε την τροπολογία 138. Ονομαστική κλίση παρακαλώ, άρχεται. Συν έναν, τον κύριο Ζήμων, υπολογίζουμε. Πέρασε. Απερίφθη. Τρία. έως 325 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 26 τραν υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 41 ήτρε υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 326 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 333 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, NV26 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 30 Ρέτζι υπέρ κατά αποχές απερίφθη 38 Τραν υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ε να βρω τη σελίδα μα το ξέρω ότι είναι η ε μετά την D αλλά τι την πήδηξα τη σελίδα για να γυρίσω πίσω ναι, βιαζόμουν και προχώρησα πολύ. Συμβαστική ε, λοιπόν, υπέρ εγκρίνεται. Συμβιβαστική F, υπέρ αποχές εγκρίνεται. G, υπέρ αποχές εγκρίνεται. H, ητά υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική I, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. J, συμβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 526 υπέρ κατά απερίφθη. 527 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβαστική και υπέρ κατά εγκρίνεται. 552 ε, τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 560 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, συμβαστική L, λάμδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, M, μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική νη υπέρ σελίδα 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική όμικρον Σελίδα 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 641 της ε, σελίδας 55, 641 τροπολογία υπέρ αποχές εγκρίνεται, συμβαστική R, ρο υπέρ αποχές εγκρίνεται 695 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 699 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική TAF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β, υπέρ κατά εγκρίνεται. 718 υπέρ εγκρίνεται. 722 υπέρ κατά απεριφθεί 115 της Ήτρα υπέρ εγκρίνεται 700 όχι συμβαστική W υπέρ εγκρίνεται συμβαστική X, χ υπερκατα αποχές, εγκρίνεται συμβαστική Y, υψηλών υπερκατα αποχές, εγκρίνεται συμβαστική Z, ζ υπέρ αποχές, εγκρίνεται και τώρα πάμε στη σελίδα 81, γυρνάμε αρκετέ σελίδες δηλαδή, και φτάνουμε στην 767 υπερκατα αποχές απερίφθη, ΑΑ συμβαστική υπέρ αποχές εγκρίνεται. 139 τροπολογία σελίδα 85 ε, υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΒ υπερκατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ αποχές εγκρίνεται. Όχι, απερίφθη, συγγνώμη. 2 ήτρε υπέρ αποχές απερίφθη. 2 τραν υπέρ όχι. Δεν καταπίπτει, δεν υιοθετηθήκε. Απερίφθη και αυτή. 32 υπερκατάποχες απερίφθη. Συμβαστική AC υπερκατάποχες εγκρίνεται. 155-156 μαζί υπερκατάποχες απερίφθησαν, 157 υπερκατάποχες απερίφθη, Τρία της Ρέτζι με τμηματική Πρώτο τμήμα υπερκατάποχες εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπερκατάποχες απερίφθη. Συμβαστική ΑΔ υπερκατάποχες εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΕ υπερκατάποχες εγκρίνεται. αφ υπερκατάποχες εγκρίνεται. ΑΓ υπερκατάποχες εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ στη σελίδα 92 είμαστε 4 υπέρ εγκρίνεται 183 υπέρ απερίφθη 184 υπέρ εγκρίνεται συμβαστική α ή υπέρ ενγκρίνεται εγκρίνεται τροπολογία 7 στη σελίδα 95 και 200 υπερκατάποχες απορρίπτονται, 199 με προφορική τροπολογία το guidance αντικαθιστά το investment guidelines υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...201 υπέρ κατά αποχές... ...201... ...στην επόμενη μας... ...κατά αποχές απερίφθη... ...και τώρα πάω στην έξι της Ρέτζη... ...υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται... 7. Όχι. Πάμε στη Ρέτζι 7. Όχι. Αλφα Ιώτα. Συμβαστική υπέρ. Σελίδα Συμβαστική ΑΙ, σελίδα 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 15 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβαστική ΑΙ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΚ υπέρ αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΛ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΑΜ υπερκατά υπέρ αποχές εγκρίνεται. 241 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 16 NV Υπερκατά αποχές απερίφθη. Ήτρε 28 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική αλφανή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλφα όμικρον υπέρ αποχές εγκρίνεται αλφα π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλφα κιού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, αΡΟ ρο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική αες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, AT υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ΑΙΟ υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται, AV υπέρ αποχές εγκρίνεται, AW υπέρ κατά εγκρίνεται. 300 υπέρ αποχές απερίφθη. Ρέτζι 16 την ψηφίσουμε και αυτήν, όχι είναι η ίδια, ΑΧ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, αλφα ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ΑΖ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ΒΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ΒΒ υπέρ υπερκατά αποχές εγκρίνεται, εγκρίνεται, BC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, BE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 323 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ονομαστικά για, την επόμ για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε, με μία ψήφο επιπλέον που θα υπολογιστεί, αρχίζει η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. The vote is closed. Πέρας. 51 ψήφοι υπέρ, 5 κατά, 52 μάλλον υπέρ η ψήφοι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους μας. Και συγχαρητήρια και στην γραμματεία, στους βοηθούς, στους ε, πολιτικούς ε, συμβούλους. Θα πάμε στην Ολομέλεια γιατί, όπως βλέπετε, ο φάκελος αυτός υπάγεται στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και άρα όλοι οι φάκελοι, όλα τα θέματα αυτά θα πάνε στην Ολομέλεια. Γι' αυτό λοιπόν δεν ζητούμε την ε, χορηγή εντολή για τη μετάβαση στους τρεις διαλόγους εδώ. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το κοινό τμήμα. Επόμενη συνεδρίαση την 3η 29 Ιανουαρίου σε, αυτό το, σε αυτή τη σύνθεση. Σας ευχαριστώ. Ήμασταν πάρα πολύ γρήγοροι και θα κάναμε ένα διάλειμμα αναγκαστικά. 9.45 έχουμε την ψηφοφορία για, την, ε, για τα benchmarks της Econ. Θέλετε να γίνει ψηφοφορία τώρα? Αν μπορεί να γίνει τώρα η ψηφοφορία. Εκτός. Φυσικά τα μέλη της Econ υποτίθεται είναι ήδη εδώ. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να κάνουμε τώρα την ψηφοφορία. Δεν ψηφίζουμε και 45, να ψηφίσουμε τώρα, αλλά χρειάζονται λίγα λεπτάκια για να φτιάξουμε λίγο τους, ε, τα μηχανήματα για την ψηφοφορία. Μια και είναι μόνο τα μέλη τη εικον. Δύο λεπτάκια διάλειμμα και μετά ψηφίζουμε.